Good afternoon, colleagues. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν συμφωνείτε, θα αρχίσουμε το δεύτερο μέρος των εργασιών μας σήμερα. Σας προτείνω να περάσουμε αμέσως στο σημείο 9. Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη ε, θα ήθελα να σας πω ότι στείλαμε μία μελή αποστολή 28 με 30 Οκτωβρίου με στόχο να επισκεφθεί η ομάδα μας, το Ινστιτούτο Καινοτοπίας Χνολογίας και της κοινότητες γνώσης και καινοτομίας της εγκαταστάσεις Βουδαπέστης και της Βιέννης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι προτείνουμε προτάθηκε από την Κομισιό ε, διατύπωση του σχετικού κανονισμού. Η κυρία Καρβάλιο, υπεύθυνη τη αντιπροσωπείας, θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό και αν θέλουν άλλοι συνάδελφοι που ήταν μέλη της αντιπροσωπείας σύντομα να κάνουν κάποια σχόλια. Θα τους δώσω το λόγο. Πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Καρβάλιο επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω θερμά μία ομάδα επισκεπτών που έχει φέρει από το Αλγάρβι, από την Νότια Πορτογαλία η κυρία Καρβάλιο. Σας καλωσορίζουμε. Έχετε τη δυνατότητα τώρα να ακούσετε την κυρία Καρβάλιο που θα μας ενημερώσει για αυτή την αποστολή. On the ITRA delegation visit in uh, Vienna and Budapest. You have the floor. Έχετε το λόγο, κυρία Καρβάλια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη και τη Βιέννη σε μία αποστολή που κατά κύριο λόγο αφορούσε την επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Είχαμε εκβαθέν συζητήσεις με του υπεύθυνου του Ινστιτούτου από το ε, διοικητικό Συμβούλιο, κάποια μέλη, τον ε, Διευθυντή, το Ινστιτούτο, άτομα τα οποία εργάζονται, ε, υπαλλήλου δηλαδή που εργάζονται στην κεντρική έδρα του Ινστιτούτου και τα ΚΙΚΣ, δηλαδή τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Τέρους, μέλη, φορείς, σε όλα τα επίπεδα συναντήσαμε και αισθανθήκαμε ότι μας καλωσόρισαν όλοι θερμά σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε ανοιχτά και εκβαθέων, πολύ ανοιχτές συζητήσεις είχαμε σε όλα τα επίπεδα με τις ε, διάφορες δομές, το Ινστιτούτο, στις κοινότητες, σε όλους τους φορείς και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους που μας συνόδευσαν, μας ξενάγησαν και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που θέσαμε. Εκτιμήσαμε όλους ιδιαίτερος αυτή την ε, επικοδομητική και ανοιχτή στάση όλων. Συλλέξαμε πάρα πολύ σημαντικές ε, πληροφορίες, γνώσεις, ε, και υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι δεν γνώριζαν πάρα πολύ καλά το Ινστιτούτο στο παρελθόν, μπόρεσαν να ενημερωθούν. Υπάρχουν δύο πολύ θετικά θέματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Πρώτα απ' όλα, με μεγάλη ευχαρίστηση διαπιστώσαμε ότι το Ινστιτούτο μπόρεσε να ξεπεράσει κάποιες διοικητικές δυσκολίες που τέθηκαν από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου το 2016. Μπορέσαμε να συζητήσουμε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα και το διοικητικό για να ρωτήσει δόθηκαν απαντήσεις και είμαστε πεπισμένοι ότι γύρισε η σελίδα, υπάρχει μια νέα επανεκκίνηση για το Ινστιτούτο πλέον. Επίσης, μας εντυπωσίασε πάρα πολύ το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που μας παρουσίαζαν διάφοροι εταίροι και οι διάφορες κοινότητες γνώσεις και καινοτομίες. Ε, πολύ λεπτομερείς παρουσιάσεις για θέματα ενεργειακά, κλιματικής αλλαγής, του τομέα της υγείας. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε λοιπόν με εκπροσώπους, με διευθυντές και όλα τα άτομα και τις επιστήμονες που μας έδειξαν τα αποτελέσματα. Είδαμε ότι υπάρχουν θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις ε, μελλοντικέ μας εκθέσεις και αυτό το συζήτησα και με την άλλη συγγετρία την κυρία Ματίας. Μεγαλύτερη διαφάνεια, άνοιγμα, καλύτερη γεωγραφική η εξισορρόπηση στην, ε, στην Ευρώπη και περισσότερη έμφαση στο τρίγωνο γνώσεων, στην εκπαίδευση. Επίσης, τα περιφερειακά κονδύλια που δίδονται μέσω των ταμείων είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ τους, ιδιαίτερως για να δημιουργηθούν συνεργίες με άλλα μέρη του προγράμματος Horizon Ευρώπης και είχαμε την εντύπωση ότι το Ινστιτούτο κατά κάποιο τρόπο είναι απομονωμένο σε σχέση με τις υπόλοιπε δραστηριότητες που λαμβάνουν η χώρα στην Επιτροπή σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία. Αυτά είναι τα κύρια θέματα. Και θα βασιστούμε σε αυτή την επίσκεψη για να ετοιμάσουμε την έκθεσή μας και τη συζήτηση που αφορούν το Ινστιτούτο Καινοτομής Τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ. Για σύντομες παρεμβάσεις τώρα θα δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Σε ένα λεπτό αν είναι δυνατόν λέει ο Πρόεδρος. Θα το εκτιμήσω. Η κυρία Λετάο Μάρκες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίδετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα κι εγώ εδώ, όπως είπε και η κυρία Γράσα Καρβάλιο, συνάδελφος, να σας πω ότι είχα την ευχαρίστηση και την δυνατότητα συμμετέχω στην επίσκεψη αυτή και θα ήθελα να πω ότι τρία πράγματα με απασχόλησαν. Πρώτα απ' όλα, η βιωσιμότητα των κοινοτήτων γνώσεων και κοινοτομίας που βρίσκονται σε μια αρχική φάση και δεν μπόρεσαν ακόμη μέχρι τώρα να βρούνε άλλα μέσα χρηματοδότησης πέραν αυτής της αρχικής περίοδου. Εάν δεν το προσέξουμε, ό,τι έκαναν θα είναι χαμένα. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε, ε, πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε κάποια χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει για τις προσεχείς κοινότητες αυτό το θέμα να το προσέξουμε και να αναπτυχθούν οι κοινότητες που υπάρχουν. Και τελικά είναι μια υπόδειξη αυτή που κάνω και όχι κριτική, να μπορέσουμε τους συντηρητές των κοινοτήτων τους θέρμισες εδώ. Είχαμε την ευκαιρία εμείς όσοι συμμετείχαμε στην επίσκεψη να τους ακούσουμε, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους και άλλες συναδέλφους για να ακούσουν κάποια πράγματα για θέματα που είναι τόσο σημαντικά για μας, οι ψηφιακές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Πεκαρίνα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω την μητρική μου, την φιλανδική. Περιμένω. Λοιπόν, εγώ δεν είχα πάει στην αποστολή αυτή στην Βουδαπέστη. και νομίζω πρώτα απ' όλα ότι είναι σαφές ότι είναι θετικό το ότι θα έχουμε κάποιες πλατφόρμες συνεργασίας ε, με εταιρείες ε, υψηλής ε, τεχνολογίας που θα έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται εντός των χωρών αλλά και στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ε, ιδρύθηκε ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη και να δημιουργήσει κάποιε ε, δυνατότητες ε, τεχνογνωσίας γιατί το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι να δημιουργήσουμε νέα εμπορικά προϊόντα. Λοιπόν, ε, δουλεύουν αρκετά καλά. Κάνουν την δουλειά που τους ανατέθηκε και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αποκέντρωση, να υπάρχει μια διοίκηση στην Βουδαπέστη, αλλά να αναλαμβάνουν δράση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, είναι κάτι που έχω σκεφτεί και εγώ άλλωστε. Γιατί αν τέτοιες πλατφόρμες θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή λύση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο τρίτος ε, πυλώνας ε, του ορίζοντα ε, συγκλίνει, αν θέλετε, με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και το ΚΙΚΣ. Ναι, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είχαμε προβλέψει πέντε λεπτά για αυτήν την συζήτηση και τα έχουμε ξεπεράσει. Αλλά υπάρχουν άλλε δύο παρεμβάσει. Από ένα λεπτό παρακαλώ. Για να πάμε στο επόμενο. Τον λόγο ο κύριο Ιζάμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να στηρίξω αυτό το οποίο είπε η κυρία Καρβάγιο. Ήμουν, ε, εγώ ήμουν στη Βιέννη και στην Πονταπέστη Συναντήσαμε εκεί πέρα επιστήμονες ε, που καινοτομούν το προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και βέβαια αυτό το οποίο με εξέπληξε είναι ακριβώς ε, το πόσο πολλοί και διάφοροι άνθρωποι ήταν. Ήταν λοιπόν μια καλή αρχή θα έλεγα. Σας ευχαριστώ. Μια που ήσταν σύντομος μπορεί να μιλήσει και η κυρία Μπάντινγκ. Στην σελίδα 4 της έκθεσης λέτε πως κάποιοι διευθύνοντες σύμβουλοι άσκησαν κριτική σε κάποιες προτάσεις. Ε, μπορείτε να επεκταθείτε ποιο ήταν το πρόβλημα δηλαδή. Ε, πρέπει να τους ρωτήσουμε τους ίδιους το τι θα έκαναν διαφορετικά από την πρόταση της Κομισιόν. Α, όλα τα ίδια είπανε. Το ένα αφορούσε την εκπαίδευση. Συμφώνησαν ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα στην εκπαίδευση, αλλά θέλουν αυτό να γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Όχι ως κάτι το ξεχωριστό. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, ανησυχούσαν για την βιωσιμότητα ακριβώ αυτού του δικτύου καινοτομία και έρευνα, ε, δηλαδή τα τρία που έχουν ξεκινήσει, κλίμα, ενέργεια και τα σχετικά, και τι θα γίνει με την σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης από πλευράς Κομισιόν και επίσης ανησυχούσαν ε, για τον προϋπολογισμό, την κατανομή του γιατί ο προϋπολογισμός ε, υποτίθεται ότι ξεκινάει μικρός και αυξάνεται. Αυτό όμω ε, δεν ισχύει για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Αυτά. Και νομίζω υπήρχαν και κάποιες παρεκκλήσεις ε, που υπήρχαν ε, στον κανονισμό και δεν υπάρχουν τώρα στην πρόταση της Κομισιόν και θα θέλαμε να τις δούμε. Και είμαι σίγουρο ότι η Μαρίζα Ματίας θα τα πει αυτά. Σας ευχαριστώ. Περνάμε εντάχει στα σημεία 10 και 11. Ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Έχουμε δύο εκθέσεις και δύο εισηγητές. Θα δώσω το λόγο και στους δύο εισηγητές για ένα πεντάλεπτο στον καθένα και κατόπιν θα ακούσουμε τους και εισηγητές για δύο λεπτά. Και όσοι είναι σκιώδης εισηγητές και στις δύο εκθέσεις θα δικαιούνται τέσσερα λεπτά. Μία ώρα και δέκα λεπτά θα ήθελα να αφιερώσουμε στο θέμα αυτό και όχι μία ώρα και 25 λεπτά όπως είχε αρχικά προβλεφθεί για να μην μείνουμε πίσω στα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινάμε με την κυρία Μαρίζα Ματίας, που είναι η συγγήτρια για, το, για την αναδιατύπωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Γκράσα Καρβάλιο για την ενημέρωση που μας έκανε της αποστολής στη Βουδαπέστη, στην οποία και εγώ συμμετείχα και φυσικά συνεργάζομαι με την κυρία Καρβάλιο. Πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια σαφή ευθυγράμμιση μεταξύ του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία και του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομία. Είναι σημαντικό να υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των δύο θεμάτων. Φυσικά δεν έχω αρκετό χρόνο για να εγγύψω σε όλα τα ζητήματα που κρίνουμε σημαντικά ε, σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού για το AID και θα ήθελα να περιοριστώ σε μερικά μόνο σημεία, να επικεντρωθώ σε αυτά για να ακούσω και τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών και των λοιπόν συναδέλφων. Έχουμε μία βασική ανησυχία που αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την τεχνική της αναδιατύπωσης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και που έχει συνέπειες όχι μόνο στη διαμόρφωση των προτάσεων, για τον κανονισμό του AID και το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομία, αλλά η μεθοδολογία της αναδιατύπωσης επηρεάζει ε, και άλλα θέματα, μια και προβλέπει μια διαχρονικότητα, μια ουδετερότητα από άποψη χρόνου. Βέβαια, ο μόνος τρόπος για να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακριβώς να ε, επικεντρωθούμε σε αυτό τη χρονική διάσταση, την διαχρονικότητα της αναδιατύπωσης. Αλλά αναφέρεται ως, η σύνδεση του κανονισμού με τα προγράμματα της Ένωσης και όχι με το ορίζον Ευρώπη. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση κατά το τέλος της, της Και αυτός είναι ένας από τους τομείς στο, στους θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ένα δεύτερο τομέα προβληματισμού αφορά το άνοιγμα και τη διαφάνεια. Ακούσαμε επανειλημμένως, ακόμη και σήμερα, στην αρχική παρουσίαση και από την Μαρία Μανουέλ, ακούσαμε το θέμα της συγκέντρωσης ε, του ΕΙΤ και των κοινοτήτων γνώση και καινοτομία. Υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση. Εμείς πιστεύουμε ότι οι κοινότητες γνώση και καινοτομία καλό θα είναι να είναι πιο ανοιχτές, πιο αποκεντρωμένες ε, και δεκτικές για περισσότερες συμπράξεις, αξιοποιώντας και τις ηχείουσες συμπράξεις και εταιρικέ σχέσεις. Να έχουμε διαφορετικά επίπεδα δηλαδή συμμετοχής, αλλά με περισσότερη αποκέντρωση και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας Τεχνολογίας και των συναφών δραστηριοτήτων. Οπότε στον κανονισμό θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια σαφή κριτήρια για την κατανομή ε, και επιβολή ε, των, επιδο των δικτών επίδοση ή το κριτήριο για τους διαγωνισμού που θα πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφανή. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το κριτήριο της αριστείας, αλλά όχι μόνο την αριστεία. Για να αποφύγουμε την υπερβολική συγκέντρωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία και Τεχνολογία. Γιατί α μην ξεχνούμε το στόχο τη της δημιουργία του AID, που είναι η πρόθεση Τη καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μείνει αναξιοποιητό το δυναμικό του AID με την υπερβολική συγκέντρωση. Άλλο θέμα αφορά τι κοινότητε γνώση και καινοτομία. Ήδη έχουμε κάποιε δραστηριότητε που δείχνουν ότι το ισχυρό μοντέλο δεν λειτουργεί απόλυτα εύρυθμα και δεν αξιοποιείται πλήρως. Γι' αυτό και θα πρέπει στον κανονισμό να προσθέσουμε κάποια μέτρα ώστε να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση και πιο αποτελεσματικός έλεγχος των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομία των ΚΙΚΣ που λέμε. Και επίσης ε, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια προθεσμία πιο σύντομη για την αξιολόγηση, για να μην ε, δεσμευόμαστε από την επταετή περίοδο αξιολόγησης που ισχύει γενικώ για το πρόγραμμα. Μου έμεινε μισό λεπτό, αλλά δείξτε λίγη υπομονή κύριε Πρόεδρε για να ολοκληρώσω. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα του προσωπικού. Γνωρίζουμε ότι στόχος είναι το ΑΕΤ να ανταποκρίνεται στα νέα κριτήρια και τις νέες απαιτήσει και προκλήσεις. Για να το κάνει όμως αυτό, χρειάζεται να είναι στελεχωμένο με το κατάλληλο προσωπικό, να έχει αρκετούς ανθρώπινους πόρους, αρκετό ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε θα πρέπει να γεφυρώσουμε τα, το νομικό κενό που υπάρχει και που απαγορεύει την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού μετά τη δεκαετία. Και ήδη θα έχουμε το πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του 2020. Και μάλιστα πριν ολοκληρώσουμε τη θητεία μας ε, δεν θα προλάβουμε να έχουμε τι διαπραγματεύσει. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια λύση με τη βοήθεια των νομικών υπηρεσιών και των διευθύνσεων ανθρωπίνων πόρων για να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει και να αποφύγουμε να χάσουμε υψηλά ειδικευμένο προσωπικό του χρόνου ή στο μέλλον, λόγω της αδυναμίας ανανέωσης των συμβάσεών τους. Αυτά είναι τα βασικά σημεία για την αναθεώρηση του κανονισμού. Φυσικά έχω κι άλλα, αλλά περιμένω με ανυπομονησία τις απόψεις και των άλλων σχεδόν εισηγητών και των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Κύρια Μαρία Καρβάλιο τώρα έχει το λόγο, που είναι η αρμόδια εισηγήτρια για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομία ε, για το 2021-2027 για την πρόθεση της καινοτομίας ε, και τη διαφύλαξη των ταλέντων στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επιλέξω κι εγώ πέντε σημεία μόνο στα οποία θα σταθώ, παρόλο που έχω ένα πολύ πιο μακροσκελή κατάλογο Παρατηρήσω και σημείων, αλλά μερικά ήδη τα ανέφερα και προηγουμένως στην ενημέρωση που σα έκανα για την αποστολή στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη. Καταρχήν, θέλουμε καλύτερη ισορροπία στο τρίγωνο της γνώσης. Να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην επιστήμη. Γιατί το ΑΕΤ στο παρελθόν ήταν πολύ συγκεκριμένο στο επιχειρηματικό σκέλος και στο σκέλος της καινοτομίας. Οπότε έμειναν αναξιοποιητές δύο πλευρές ε, του τριγώνου, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ε, που περιλαμβάνονται ήδη στις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, ε, μεταπτυχιακές σπουδές στο ψηφιακό κόσμο ή στον επιχειρηματικό κόσμο, επαγγελματική κατάρτιση, αλλά σε σχέση με τη βασική δραστηριότητα της κάθε κοινότητας γνώσης και καινοτομίας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που θέλουμε να προτείνουμε ως αλλαγή στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο σημείο που με βρίσκει σύμφωνη με αυτά που είπε η κυρία Ματίας αφορά το άνοιγμα και τη διαφάνεια οι πρώτοι διαγωνισμοί, οι πρώτε προσκλήσεις για υποβολή προσφορών ήταν πολύ διαφανεί από το ΕΤ. Στη συνέχεια όμως, και όταν δημιουργήθηκαν νέε κοινότητε γνώση και καινοτομία ε, και επεκτάθηκαν οι συμπράξει σε νέους εταίρου, μερικοί αντιτάχθηκαν κατά των ανοιχτών και διαφανών διαγωνισμών. Θα θέλαμε λοιπόν να μεριμνήσουμε να είναι οι ανοιχτές οι προσκλήσει για υποβολή προσφορών και προσιτές προς το φάσμα εταίρων για συμπράξει. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική εξισορρόπηση, εκεί έχω κάποια διαφορά και διαφωνία με τη Μαρίζα. Εγώ θεωρώ ότι η αριστεία θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια γεωγραφική ισορροπία, ακόμη και με το κριτήριο της αριστείας ώστε να βρούμε τους μικρούς θύλακες αριστείας που υπάρχουν παντού στην Ευρώπη. Και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θέλουμε πιο γεωγραφικά ισορροπημένη κατανομή των κοινοτήτων γνώση και καινοτομία, κρατώντας όμως την αριστεία ως το βασικό κριτήριο. Όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας. Γιατί δυστυχώς η κατανομή ε, επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε μερικές περιφέρειες και έχουμε συγκέντρωση στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το, τα περιφερειακά κονδύλια του AID και να βρούμε έναν σωστό κατάλληλο τρόπο ώστε το AID να συνεργάζεται με το ή καθόλο καθόλου, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Και το συζητήσαμε αυτό με το ΑΙΤ αλλά και με το AIC. Και το αναφέρουμε στην έκθεση. Θα πρέπει να φροντίσουμε για περισσότερη συνεργασία μεταξύ των δύο του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομίας του ΑΙΚ δηλαδή. Επίσης, είναι κρίμα που δεν έχουμε μια σταδιακή μείωση ε, των ε, δραστηριο... της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων που απομακρύνονται από την αγορά και να μην χάσουμε τη γνώση και την εμπειρία που ήδη έχει δημιουργηθεί. Θα πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη χρηματοδότηση στις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, στις ΚΙΚΣ. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι για τις δύο νέες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Η πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για δύο νέες και προτείνει ως πρώτο θέμα είναι οι δημιουργικές βιομηχανίες. Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή, αλλά αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της, του θέματος για τη δεύτερη κοινότητα γνώση και καινοτομία. Και υπάρχει μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει κάνει μελέτη αντικτύπου για πολλά θέματα και ένα από τα θέματα αυτά που καλύπτονται από τη μελέτη αντικτύπου είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και θα θέλαμε να το σκεφτούμε με τους και ηγητές και τους α, συναδέλφους. Για μας είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για όλη την Ευρώπη και να μην πω για τον κόσμο. Και δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με το θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνόλογης και αφορά το είδωρ την λειψιδρία, την ποιότητα του νερού, σε όλους τους υδάτινους, όλες τις υδάτινες λεκάνες, ποτάμια, λίμνες, ωκεανούς, γιατί έχουμε καινοτομίες γνώση και καινοτομίες για τα τρόφιμα, για την ενέργεια, την υγεία, το κλίμα, αλλά για το νερό δεν έχουμε καμία, γιατί λοιπόν η δεύτερη νέα κοινότητα γνώση και καινοτομίας να μην αφορά το νερό. Αυτή είναι μια πρόταση που καταθέτω στο τραπέζι για να τη συζητήσω με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ κυρία Καρβάλιο και τώρα να ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές για την έκθεση κυρίας Μαρίζα Ματίας πρώτα. Ο κύριος Άντρης Κουμπίλιος είναι ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Η έκθεση αυτή για τον κανονισμό είναι πιο εύκολη από αυτό το θέμα της στρατηγικής για το Ινστιτούτο. Το ερώτημα όμως είναι πώς βλέπουμε την όλη στρατηγική για το μέλλον αρκεί αυτό που προτείνει στον κανονισμό στην αντιτύπωση η Κομισιό. Υπάρχουν διάφορα θέματα εκτός από αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Δεκαρβάλιο και δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε στον κανονισμό απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Προσπαθώ να κατανοήσω κάποια πράγματα, τι ακριβώς κάνει επίσης και το Ινστιτούτο και για μένα η πιο σημαντική του αποστολή ολοκληρώθηκε με την ίδρυση των ΚΙΚΣ αυτών των κοινοτήτων. Μήπως πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε και κάποιες ομοδοποίησεις, κάποια κλάστερ, μήπως ό,τι έγινε εκεί θα πρέπει να γίνει και σε άλλες χώρες, σε όλες τις ε, σε όλους τους πυλώνες, σε όλους τους τομείς. Τώρα είναι θέμα ε, μόνο καινοτομίας μόνο εκπαίδευσης. Πού αποφασίζονται όλα αυτά τα οποία γίνονται πραγματικότητα στην καινοτομία. Στη Silicon Valley πολλές φορές το βράδυ σε ένα μπαράκι, σε ένα pub, σε ένα ποτό αποφασίζονται και τα κάποια πράγματα. Εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πού μπορούν να συμβούν αυτά. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, εάν το Ινστιτούτ πρώτα απ' όλα αφιερώνει το έργο του στη δημιουργία των κοινοτήτων και μπορούν να βοηθήσουν startups ή στην εκπαίδευση. Είμαστε τώρα σε μία περίοδο κατά την οποία οι πρώτες αυτές κοινότητες θα πρέπει να έχουν βεβαίως και μία οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να επιβιώσουν από ό,τι κατάλαβα πρέπει να απαντήσουν σε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Ερώτημα λοιπόν στρατηγικής. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολή του Ινστιτούτου για την δημιουργία των κοινοτήτων ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν βιώσιμο, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι δεν επιβιώνουν ή δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν οι κοινότητες. Αν δούμε επίσης ε, για τα κλάστερ την βιβλιογραφία, βλέπουμε ότι τα συμπεράσματα είναι ότι αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργηθεί δηλαδή μια διοικητική δομή σε πρώτη φάση, γιατί δεν επιβιώνουν αν δεν προχωρήσουν περισσότερο. Και το ερώτημα είναι, το Ινστιτούτο πραγματικά παράγει αυτό το οποίο ε, δημιουργήθηκε, δηλαδή τα περίφημα αυτά κλάστερ, αυτές τις κοινότητες για να ενεργήσουν στους ε, τομείς αρμοδιότητες ή μήπως αυτές οι κοινότητες δεν ενδιαφέρουν, δεν ενδιαφέρουν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό. Αν δούμε τι γίνεται με την καινοτομία ή μέσω μικρών επιχειρήσεων ή κοινοτήτων ή μεγάλων επιχειρήσεων. Έχουμε, είχαμε την Nokia, τη Siemens, που άρχισαν πριν από χρόνια να είναι καινοτόμε και ίσως μετά εξαφανίστηκαν. Το Ινστιτούτο θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικό και προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διότι χωρίς την δική τους υποστήριξη η καινοτομία δεν μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές για τις δύο εκθέσεις έχουμε την κυρία Γκαλβές Μουνιός. Θα μιλήσω ισπανικά τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συναδέλφους Καρβάιο και Ματίας για τη θέση του. Συμμεριζόμαστε τα περισσότερες ε, ερωτήσεις που τέθηκαν και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν. Πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσουμε καλύτερα την ε, ε, ισορροπία σε αυτό το τρίγωνο των γνώσεων, ενίσχυση, εκπαίδευση, της επιστήμης και καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, δεδομένου ότι ειδικά είναι, δεν είναι ισοσκελισμένο το θέμα αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα και με τις συναδέλφους ότι η αριστεία θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο κατανομής, αλλά βεβαίως θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να δούμε πρωτοβουλίες πιο συμπεριληπτικές και λαμβάνοντας υπόψη και σε περιφερειακό επίπεδο τις διάφορες σε διάφορες περιφέρειες και περιοχές. Υπάρχουν χώρες που χρειάζονται ειδική προσοχή, ενώ άλλες περιοχές της Ευρώπης στην, ε, στα κράτη μας δεν το χρειάζονται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ πύκνο κατοικημένες περιοχές που δεν ε, εκπροσωπούνται, που δεν έχουν καμία τέτοιου είδους κοινότητα γνώσης και καινοτομίας. Τρίτο στοιχείο ισορροπίας. Το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Τι σημαίνει αυτό. Ότι στο Ινστιτούτο, στο οποίο υπάρχουν πρωτοβουλίες για να διορθωθεί το θέμα αυτό, υπάρχουν ακόμη ανισορροπίες. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Ματίας ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το πρόβλημα το εργασιακό που υπάρχει στο Ινστιτούτο. Και αν θέλουμε να του αναθέσουμε περισσότερα καθήκοντα για να αναπτυχθεί περισσότερο και να αυξήσει τις δραστηριότητες, θα χρειαστεί περισσότερο προσωπικό. Άρα δεν είναι λογικό να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τα πιο έμπειρα άτομα που εργάζονται εκεί. Θα πρέπει να αναζητηθεί λύση λοιπόν, διότι δεν μπορούμε να τα χάσουμε αυτά τα άτομα. Δεν είναι καλό ούτε για το Ινστιτούτο, ούτε για τις κοινότητες, ούτε γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι όλε οι κοινότητε δεν είναι ίδιε. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι δεν βρίσκονται στην ίδια θέση. Βεβαίω άλλε άρχισαν πριν, έγιναν, ήταν περισσότερο εμπειρική η πολιτική για, με τι πρώτε από ό,τι για τι μεταγενέστερε. αλλά δεν βρίσκονται όλες στον ίδιο τομέα και δεν έχουν όλες την ίδια δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων ισότιμα. Υπάρχουν τομείς που είναι πιο ελκυστικοί άλλους. Αυτή λοιπόν η ποικιλομορφία που υπάρχει θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τελικά θα ήθελα να αναφερθώ και στις νέες κοινότητες. Το IRC, το HSC έκανε το Κοινό Ινστιτούτο Ερεύνων έκανε μία έκθεση για τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτές οι νέες κοινότητες και αυτές οι οποίες αφορούν τα είδα του τους ωκεανούς είναι ενδιαφέροντες δεδομένου ότι υπάρχουν στο Horizon Europe και άλλους τέτοιες, και άλλους τέτοιες πρωτοβουλίες. Ίσως να υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, άλλες περιοχές της Ευρώπης που να μην είναι ε, πάρα πολύ καινοτόμε σε άλλους αλλά έχουμε να κάνουμε εδώ και με την κοινωνική ε, καινοτομία, αν μπορούσα να το πω. Συμπερίληψη, ε, μεταναστευτικό Άρα ο τομέας αυτός θα μπορούσε να είναι από τους επόμενους τομείς του οποίου θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που ήθελα να πω και να συμφωνήσω με τι συναδέλφου ότι όντω ε, είναι κάπως απομονωμένο φαίνεται το Ινστιτούτο αυτό από την γενική στρατηγική καινοτομία και θα πρέπει κάτι να κάνουμε σοβαρά για να μπορέσουμε να βρούμε συνέργειες. Έχουμε ένα μέσο στη διάθεσή μας πολύ σημαντικό αλλά θα πρέπει να μάθουμε να το εκμεταλλευόμαστε θετικά καλύτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ίζαψ, εκ μέρους της, ε, εκ μέρους της κυρίας ε, Σολής Παρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την στήριξή μου στο έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, αλλά κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θα ήθελε η ομάδα μας. Πρώτα απ' όλα το θέμα αυτό που λέτε του να είναι ανοιχτό αυτό το και γνώση και καινοτομίες. Ξέρουμε βέβαια ότι ε, υπάρχει μεγάλη αυτή αυτονομία και μπορεί το Ινστιτούτο Τεχνολογίας να δημιουργεί νέες τέτοιες κοινότητες. Αν είναι να προχωράμε προς τα εμπρό και ο βασικός στόχος είναι να παράγει ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον καινοτομία, τότε το να είναι πιο ε, ανοιχτέ αυτές οι κοινότητες ε, έχει μεγάλη σημασία και αυτό αφορά ακριβώς και το ότι θα πρέπει να φαίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, μιλάμε με κάποιους ε, συναδέλφους μας και μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, αρκετοί από εμά ε, δεν ξέρουν τι είναι. Παρά το ότι είναι ένα έργο το οποίο υπάρχει ήδη εδώ και 11 χρόνια. Βεβαίω είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί μέσω των ε, κόμβων αυτών καινοτομίας στα κράτη-μέλη. Η δεύτερη ερώτηση βεβαίως αφορά την ε, γεωγραφική εξάπλωση. Συμφωνώ με τα κριτήρια αριστείας, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον καινοτομία, αλλά και χώριο στα κράτη-μέλη. Υπ' αυτήν την έννοια το έργο αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και από εθελοντικό να γίνει υποχρεωτικό. 10% σύμφωνα με την πρόταση της ε, Κομισιόν ε, θα αφιερωθεί στο περιφερειακό αυτό σχέδιο. Κατά την άποψή μου μπορεί να είναι και περισσότερο. Και το τρίτο θέμα που ανέφεραν ήδη κάποιοι συνάδελφοι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των ε, κοινοτήτων. η ότι υπάρχει σταδιακή κατάργηση και ότι υπάρχει παρακολούθηση πιο συχνή μετά από τα 7 έτη είναι πάρα πολύ καλή. Το σκεπτικό είναι να υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και μετά από το 15ο έτος και αυτό ήταν ακριβώς το νόημα του μνημονίου. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει και πρέπει νομίζω να βάλουμε στην ατζέντα της καινοτομίας ε, λίγα περισσότερα πράγματα του τι σημαίνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όσον αφορά δε το τελευταίο, τις νέες τέτοιες ε, κοινότητες, ε, μία από αυτές έχει ήδη προταθεί Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, Μιλάμε για το 10ο έτος, το 2025. Καλό είναι να υπάρχει μια διαφάνεια για το πώς δημιουργούνται αυτές οι νέες κοινότητες. Είτε μιλάμε για το νερό, είτε αφορά τη μετανάστευση που επίσης έχει αναφερθεί. Οπότε η διαφάνεια νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ για τους ε, πράσινους. Έχουμε τον ίδιο σκιώδη και για τα δύο θέματα, τον κύριο Μπούχνερ και του δίνω τον λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θεωρώ ότι η δουλειά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν ελλείμματα στην δομή της έρευνας ε, και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και το περιβάλλον, το δημιουργικό. Γι' αυτό είναι νομίζω αποφασιστικό για την καινοτομία μας ε, τις επόμενες ε, δεκαετίες, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος προϋπολογισμός. Και εδώ πέρα ήδη τα είπαν και άλλοι προλαλήσαντες, ότι χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Έχω προβλήματα επίσης με την ε, θεσμική συνεργασία και τον ορίζοντα. Δεν έχω πιστεί ότι αυτό ανταποκρίνεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των κοινοτήτων αυτών. Ένα παράδειγμα. Η προϋπόθεση του 40% των κρατών μελών που θα πρέπει να είναι σε μια συνεργασία. Σε κάποιους τομείς έχει νόημα, αλλά όχι σε όλους. Εγώ ο ίδιος ήμουν διευθυντής μιας ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας στον τομέα της έρευνας ε, και αυτοί οι περιορισμοί συχνά είναι πάρα πολύ ε, δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα κριτήρια επιλογής για τις νέες αυτές κοινότητες, τα οποία πρέπει να είναι σαφή και με διαφάνεια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και βεβαίως πρέπει να γίνει μια επιλογή, αλλά θα πρέπει η επιλογή αυτή να έχει την μορφή της μεγαλύτερης δυνατής ε, διαφάνειας. έτσι ώστε αυτές οι κοινότητες να μην είναι κλειστές λέσχες αλλά να μπορούν να γίνουν δεκτοί και νέοι εταίροι. Αυτό ισχύει ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, δεν έχουν υποχρεωτικά όλες τις ε, νέες ε, πληροφορίες των ιδρυτών νέα κέντρα αριστείας σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν αρκετή καινοτομία είναι οπωσδήποτε αρκετά σημαντικά αλλά το τόνισαν και αυτό οι προλαλήσαντες. Η αριστεία είναι ακόμα σημαντικότερη. Πολύ απλά για κάποια θέματα κάποιες περιφέρειες έχουν καλύτερες προοπτικές και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Οπότε να πούμε ότι όλη η Ευρώπη έχει ένα σύστημα ή να έχουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένο ποσοστό δεν είναι σωστό. Και τέλος. Έχουμε μεγάλες ε, δυσκολίες για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει οι ίδιοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι στόχοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν στην αποστολή και στους στόχους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, ειδικά στην ε, στρατηγική της ε, καινοτομίας. Θα πρέπει δηλαδή οι αρχές της ε, αηφορίας να λαμβάνονται υπόψη στα επιχειρησιακά σχέδια. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και τώρα για την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία έχουμε δύο σκιώδεις ηγητές. Δύο λεπτά το πολύ ο καθένας παρακαλώ. Ο κύριος Ανδρέα Καρόπο είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, μίλησα πιο πριν, ε, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρβάλιο που ήταν επικεφαλής ε, στην ε, Βουδαπέστη. Πραγματικά τρέχαμε χωρίς ούτε ένα λεπτό ξεκούρασης. Ε, συνεχώς ε, δουλεύαμε μια εξαιρετική αποστολή και χάρη στην δουλειά που έκανε η Επιτροπή. Κάποια πράγματα τώρα για τα συγκεκριμένα θέματα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην ανάλυση που έχει γίνει για το Ινστιτούτο αυτό υπό την έννοια την εξής τα ε, follow-up ε, τα οποία έχουν δοθεί από το EIT απαντάνε στην κριτική της ε, Κομισιόν. Γιατί, όπως έλεγε και ο κύριος Μπούχνερ, έχουμε εδώ πέρα έναν κάπως κλειστό κύκλο, ένα κλειστό κλαμπ, κάπως πιο απομακρυσμένο σε θέματα δηλαδή διαφάνειας Τώρα, για το θέμα του εάν είναι ορατό. Ε, κοιτάξτε, το ακούει κανείς και έχει την εντύπωση ότι είναι μια, κάτι το συγκεκριμένο, ένα, κάτι το σταθερό και όχι το δυναμικό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το όνομα γιατί και κάποιος άλλος το είπε. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μας ε, με τους οποίους μιλάμε εδώ πέρα δεν ξέρουν ε, περί τίνος πρόκειται. Φανταστείτε τι συμβαίνει ε, παραπέρα στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, να φανταστούμε λοιπόν κάτι το οποίο θα είναι πιο αντιληπτό αμέσως ότι αποτελεί μια κοινότητα. Και μετά βεβαίως υπάρχει και η σχέση αυτή που ανέφερε και ο κύριος Πακέ. Το Horizon πηγαίνει προς ε, μια διακλαδικότητα εγκαταλείπτει τις δέσμες ενώ εμείς ακολουθούμε έναν δρόμο διαφορετικό ειδικά επίσης ε, και για τον κλάδο τον δημιουργικό και τον πολιτισμικό έχουμε νομίζω φύγει τελείως από τα όσα γίνονται στο νέο πρόγραμμα Horizon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα... Πάμε στο δεύτερο σκιώδη γιατί της ομάδας ε, Ταυτότητας και Δημοκρατίας, την κυρία Ελένα Ρίτσι. Ευχαριστώ την παρουσίαση της έκθεσης για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας. Ω εκπρόσωπο τη ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήμασταν ανέκαθεν υπέρ τη έρευνα και τη καινοτομία, εφόσον φυσικά αποφέρουν η έρευνα και η καινοτομία απτά ωφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Βέβαια, ε, το, το Τμήμα Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, υπογραμμίζει σχετικά με την έρευνα αντικτύπου ότι 73% των κονδυλίων του ΑΕΤ ε, συγκεντρώνεται σε πέντε χώρες μόνο. Στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την ε, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν έχουμε αρκετή ολοκλήρωση και πρόωθηση των ε, δραστηριοτήτων των κοινωτών γνώσεων και καινοτομία σε όλη την Ευρώπη. Άρα είναι περιορισμένο ο αντίκτυπό του. Επίση, η πρόταση θέλει να ενισχύσει τα, την καινοτομία χωρί να προβλέπει όμω με ποιου τρόπου, με ποια συγκεκριμένα και αυτά μέτρα και με βάση ποιε παραμέτρου. Πώς πρόκειται λοιπόν να δημιουργήσουμε καλύτερη ισορροπία των πόρων μεταξύ των κρατών μελών για να αποφευθεί η συγκέντρωση, όπως ρώτησε και οι προελαλήσαντες. Επίσης, το, στη μελέτη αντικτύπου που έστειλε πριν την 1η Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται ότι το 73% των ανοιχτών διαβουλεύσεων καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητε τη τριτοβάθμιας εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα δεν περιλαμβάνονται παρκώς στα περιφερειακά και τοπικά οικοσυστήματα. Οπότε, πότε θέλε, πώς προτίθεστε να αποκαταστήσετε αυτές τις ανισορροπίες. το κόμμα μου η Λέγκα θέλει να προωθήσει τη διαφάνεια των κοινοτήτων γνώση και καινοτομία για να έχουν θετική έκβαση τα σχέδια και προγράμματα και να έχουν τοπική προστιθέμενη αξία. Στο ίδιο όμως, έγγραφο αναφέρεται σε ένα υποσημείωμα της, υποσημείωση της σελίδας 53 ότι κάποιες κοινότητες γνώσης και καινοτομία εξέφρασαν την απογοήτευσή τους γιατί δεν έχουν αρκετούς ε, εταίρους και γιατί υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση των κονδυλίων. Και αυτό είναι πρόβλημα και δημιουργεί ανισορροπία. Πώς προτεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και να εξασφαλίσει μια διαφάνεια στην κατανομή των κονδυλίων. Σε τι θα δώσετε προτεραιότητα, στην αριστεία ή στη γεωγραφική ανακατανομή. Επίσης, ε, λάβατε υπόψη ανησυχίες των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Έγιναν ε, έλεγχοι. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θέλει να αυξήσει τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της ε, έρευνας προκειμένου να ε, εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές ταλέντων. Είμαστε υπέρ τέτοιων συμπράξεων και δραστηριοτήτων και θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί μερικές φορές ε, παραγωνίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη διαδικασία αυτή λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Επίσης, ε, ε, τι γίνεται με ε, το, το σήμα 8 σε μερικές μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται αυτό το Ινστιτούτο θα θέλαμε όχι μόνο τα έγκυρα και φημισμένα πανεπιστήμια να είναι επιλέξιμα για κονδύλια και να προτείνουν προγράμματα. Θα πρέπει και μικρότερες κλίμακες πανεπιστήμια να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για προγράμματα, για να έχουμε μια πιο εξισορροπημένη γεωγραφική κατανομή και πιο απτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη διανομή αυτού του σήματος του AID. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του ECR έχουμε τον ίδιο σκιώδη συγητή που ασχολείται και με τις δύο εκθέσεις. Ο κύριος Ρόμπρους, που αντικαθίσταται όμως από τον συνάδελφο τον κύριο Ρόκαν. Ευχαριστώ. Δυστυχώς, κύριε Ρούς, ε, είναι σε αποστολή στην Ουάσιγκτον. Ο κύριος μάλλον ε, ε, θα ήθελα να σας μεταφέρω τα έξω σχόλια του αρμοδίου για του θα πρέπει να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άγχος που δημιουργεί πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην έρευνα. Υπάρχουν κοινότητε γνώση και καινοτομίε που τα πάνε καλά και άλλε ε, που έχουν προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Οπότε ρωτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ έχει κατάσταση σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία θα πρέπει να δημιουργήσει αυτό το τρίγωνο τη γνώση, όπω ε, είπαν οι προλαλήσαντες. Και δεν ξέρω σε, ποιο, σε ποια πλευρά του τριγώνου θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση, στην αγορά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αγορά. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική ισορροπία, ο Μπάς εμ, θεωρεί ότι το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η αριστεία. Σε ό,τι αφορά τι συνέργειες με το Horizon Ευρώπη, συμφωνεί ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε συνεργασίες και συνέργειες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καινοτομία. το Πώ Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αποφύγει αυτέ τι επικαλύψει σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα. Ε, φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε τις κοινότητες που δεν είναι ακόμη βιώσιμες, αλλά για μια περιορισμένη μεταβατική περίοδο. Και αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται υπό όρους. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας που δεν είναι αποτελεσματικές. Ο κύριος Ρούς προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους και και φυσικά με τις εισηγήτριες. Μάλιστα. Η κυρία Μαρίζα Ματίας είναι η σκιώδη συγκίτρια της ΓΚΟΕ για το δεύτερο θέμα, την έκθεση της κυρίας Καρβάλιο. Ε, θέλετε τώρα το λόγο ή μετά όταν θα δευτερολογήσετε για τη δική σας έκθεση. Αργότερα, λέει η κυρία Ματίας. Καλώς. Τρεις άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Έλερ πρώτος. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ας μην ξεχνούμε τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο πιο διεξοδικά. Αν δούμε τις στατιστικές σε σχέση με τη γεωγραφική ισορροπία, κρίνουμε εύκολο ότι υπάρχει συγκέντρωση σε πέντε χώρες. Αν όμως δούμε τους κόμβους, το τοπίο αλλάζει, η εικόνα που αποκομίζουμε είναι διαφορετική. Οπότε είναι δύσκολο να διαμορφώσουμε το θεματολόγιο του ΑΕΤ και να το επικεντρώσουμε σε πιο στερημένες περιοχές, γιατί το, ο μηχανισμός των κόμβων είναι το πιο σημαντικό και πιο αποτελεσματικό, γιατί μπορούμε να βρούμε κάποιες περιοχές που υστερούν, αλλά που έχουν πρόσβαση στους κόμβους. Θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων Αυτά τα εκπροσωπούν πολλέ φορέ οι κοινότητε γνώση και καινοτομία. Το θέμα είναι πώς θα γίνει καλύτερη διάδοση. Γιατί να μην εξετάσουμε περισσότερο τα hubs, τους κόμβου. Μπορεί να έχουμε επικρίσεις για τους κόμβους, αλλά αν επικεντρωθούμε μόνο στη στατιστική συγκέντρωση των ΚΙΚΣ, ε, είναι παραπλανητική η εικόνα που δημιουργείται. Και οι... ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, είναι από τα πανεπιστήμια. Αλλά πολύ συχνά δεν έχουμε αρκετέ γυναίκε σε επιστημονικέ σπουδέ ή στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό για να αποκαταστήσουμε μια μεγαλύτερη ισορροπία των φύλων, αλλά οι κοινότητε εξαρτώνται από του συμμετέχοντε που προέρχονται από τα πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμεί ποιο θα προέλθει από τα πανεπιστήμια και δεν έχουμε αρκετέ γυναίκε εκεί. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τη βιομηχανία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον πολιτικό χαρακτήρα της απόφασης. Γιατί θεωρήσαμε το κλίμα και την ενεργειακή καινοτομία σημαντικούς τομείς για τις κοινότητες. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουμε αρκετούς, αρκετούς επιχειρηματίες, γιατί θέλουμε να προωθήσουμε τη μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Εκεί δεν υπήρχε ένα επιχειρηματικό αντίβαρο και ένα εργαλείο στην αγορά, ένας μηχανισμός της αγοράς. Γιατί αν έχουμε μια κίκη για το κλίμα, συζητήσιμο βέβαια, καλώς, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι την αρχή το δημιουργήσαμε με ένα ευχολόγιο και έτσι απομακρυνθήκαμε από την αρχική ιδέα του τριγώνου τη γνώσης και η προσπάθεια να τροποποιήσουμε την εκπαίδευση ώστε να διαφερθεί περισσότερο για την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια κοινότητα νεοφιών επιχειρήσεων με μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα καινοτομίας. Ίσως η καλύτερη πηξίδα α, μας θα πρέπει να είναι η έκθεση του ενεκτικού συνεδρίου. Γιατί έγιναν πολλές εκθέσεις και μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια και αν ανταποκρίνονται ε, στον ορισμό που έχουμε δώσει για την επιτυχία. Το θέμα είναι, είναι σωστός ο ορισμός μας για την επιτυχία. Και αυτό που έδειξε το ελεκτικό συνέδριο είναι η σωστή κατεύθυνση, γιατί πρώτη φορά έγινε έλεγχος με μια πρόπτικη και αντικτύπου. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ καλή πηξίδα η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για τα μελλοντικά επιτεύγματα που θα ζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης δεν μπορούμε να υπερφορτώνουμε αυτό το μηχανισμό. Και το επιχείρημα ότι δεν έχει πανευρωπαϊκό αποτέλεσμα, αρχικά το AID θέλαμε να γίνει το Ευρωπαϊκό MIT. Και τώρα είπαμε καλά, ας επικεντρωθούμε στην αρχή με σε ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία με λίγε κοινότητε γνώμη και καινοτομία, γιατί δεν μπορούμε με ένα προπολογισμό τριών δισεκατομμυρίων να αλλάξουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και να την κατευθύνουμε περισσότερο προ την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με πέντε μόνο κικ, με πέντε μόνο κοινότητε γνώση και καινοτομία. Αυτέ οι λίγε κοινότητε γνώση και καινοτομία είναι το σημείο αφετηρία. Αλλά νομίζω ότι η πολύ επικριτική και ε, οξυδερκή έκθεση ήταν αυτή το ελεκτικού συνεδρίου που μπορεί να μας κατευθύνει και στη συνέχεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μόνο μία ποσοτική απαρίθμηση των ορών που αφιερώθηκαν, αλλά να δούμε τι μέλλον θέλουμε για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Ευχαριστούμε κύριε Έλερ. Κύριε Λετάου Μάρκε. έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να υπογραμμίσω τρία θέματα που μου φαίνονται σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, το Ινστιτούτο και οι κοινότητε δημιουργήθηκαν να λύσουν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή να περάσουμε από τα αποτελέσματα τη έρευνα στην καινοτομία. Το είχε η Ευρώπη αυτό το πρόβλημα και συνεχίζει να το έχει. Η Ευρώπη εννοώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, το θέμα αυτό θα πρέπει να το επιλύσουμε. Εγώ ομολογώ ότι δεν γνωρίζω, αλλά ίσως κάνω λάθος, πολλές περιοχές και χώρες του κόσμου, στις οποίες τέτοιου είδους προβλήματα επιλύονται χωρίς μία δημόσια βοήθεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι μια τέτοια βοήθεια δεν μπορεί να είναι αιώνια, αλλά δίνει την απαραίτητη όθηση. Και αυτό είναι αυτό που θέλω να υπογραμμίσω. Και αυτή είναι η θέση των σοσιαλιστών. Δεύτερον, όταν μιλούμε για βιωσιμότητα αυτών των κοινοτήτων, δεν θέλουμε να πούμε ότι η παρούσα προστιθέμενη αξία των πρώτων δεν είναι κάτι το ορατό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν εδώ επιχειρήσεις ή άτομα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία σε διάφορους τομείς της ενέργειας Φερρυπίν για να μας πούνε κάποια πράγματα όπως εμείς πήγαμε εκεί και είδαμε περί τίνος πρόκειται. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και τελικά δεν συμμερίζομαι την ιδέα ε, που ε, χρησιμοποιούν κάποιοι. Αχ, τις καημένες, τις μη ευνοημένες περιοχές. Ακούστε, εμείς ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν εξαιρετικοί ερευνητές, υπάρχει αριστεία και υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν όλα αυτά τα κριτήρια. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κάτι τέτοιο να συνεχιστεί να υπάρχει ως διαθέσιμο υλικό και προσωπικό μόνο σε μερικές περιοχές της Ευρώπης και όχι σε όλες. Θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπάντιν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Λαμβάνε εδώ συγγήτρια γνωμοδότησης εκ μέρους της Κούλτ από εκπαιδευτικής πλευράς. Ας πω κάποια θέματα. Επίσης πρέπει να πω ότι έχω κατά νου και κάποια θέματα που αφορούν και την Ήτρε. Κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το επίπεδο φιλοδοξιών, έτσι όπως ε, το προβλέπει η νομοθεσία. Πολύ με ανησύχησαν αυτά που διάβασε η νομοθεσία, διότι πραγματικά δεν μιλάει καθόλου για φιλοδοξία και πολύ λίγο για επιστήμη καινοτομία. Ε, μετά από αυτά τα οποία άκουσα με τον διευθυντή του ΣΑΙΤΗ, ότι η ποιότητα είναι καλή, υπάρχει ε, πραγματικά φιλοδοξία και θα ήθελα αυτό να προβλεφθεί και στην νομοθεσία. Ε, αν δεν μπορέσει κανείς να εφεύρει, να ανακαλύψει νέα πράγματα, τι είδους καινοτομία κάνει. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Πρόκειται για Ινστιτούτο καινοτομία και Τεχνολογίας. Δεν πουλάμε μόνο ιδέε ε, στη θεωρία, αλλά στην πράξη ιδέε που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Τώρα, αν δούμε τώρα πώς μπορούν να επεκταθούν και να πάνε παντού ε, ε οι δραστηριότητε αυτού του Ινστιτούτου. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ανάγκη ανώτατη εκπαίδευση υψηλών επίπεδου στάνταρ και φιλοδοξιών. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και νομίζω ότι στα μεταξύ των μελών IRS ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ποσοστά και των κονδυλίων του προπολισμού που προβλέπονται, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι στις χώρες IRS και για την επιχειρηματικότητα. Ακούστε, έχουμε λαμπρά μυαλά και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Εξίσου. Το σύστημα το εκπαιδευτικό είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να είναι προσβάσιμο σε όλους. Έχοντας αυτά κατά για την χρηματοδότηση, μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικό το νέο πρότυπο. Ε, υπάρχουν ίσως κάποιες ανησυχίες, αλλά θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον 30% των ευθυνών του ε, Ινστιτούτου και των Κοινοτήτων είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια κερδοφόρος δραστηριότητα. Θέλουμε λοιπόν ε, να μπορέσει να αναπτυχθεί κάθε κοινότητα και να αυτοχρηματοδοτείται, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να το ισοσκελίσουμε με την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ε, η έρευνα μπορεί να αποφέρει χρήματα μόνο όταν είναι καινοτόμα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ, ε, και να ξέρουμε ότι πρόκειται οι κοινότητες ανεξάρτητες. Επίσης, δεν θα πρέπει να πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα. Τώρα όσον αφορά την ορατότητα. Πριν έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν μου δόθηκε αυτός ο φάκελος δεν είχα ακούσει το θέμα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν ε, ε, υπεύθυνη δημοσιογραφία επιστημονικά θέματα και δεν ήξερα τίποτα για αυτά τα θέματα. Αυτό πραγματικά είναι τρομερό. Και τώρα βλέπω πόσο Μεγάλη ποιότητα έρευνα γίνεται, αλλά πρέπει να πω ότι σε θέματα διαφήμιση κατά κάποιο τρόπο και ορατότητος δεν είχε γίνει τίποτε. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν η κοινή γνώμη γενικότερα θα είναι πιο καλά ενημερωμένη, όταν μάθουν όλοι ότι υπάρχει, θα ενημερωθούν έγκαιρα και θα μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσει. Τώρα, εάν θέλουν να Θέλουμε να συνεχίσουμε όλα αυτά, οι άνθρωποι από αυτά τα όργανα να τους υποστηρίζουμε, οι υπεύθυνοι. Θα πρέπει να έρθουμε εδώ, να οργανώσουμε μια ακρόαση, να γίνει γνωστό τι κάνουν για να τους υποστηρίζουν καλύτερα. Όσον αφορά τώρα στην πρόταση για CCI, και την αρχή του εκ μέρους Επιτροπής Πολιτισμού δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Ινστιτούτο Καινοτομίας Τεχνολογίας και τα περισσότερα έσοδα τουλάχιστον σήμερα σε αυτήν τις νέες τεχνολογίες προέρχονται από το κινηματογράφο, από τα έσοδα του ίντερνετ, από το ε, απευθείας μετάδοση, το Ηνωμένο ε, Βασίλειο όπως ε, ξέρετε, έχει τις περίφημες μέσα που όπως λέγεται, είναι, ονομάζονται Harry Potter. Πρέπει να πω ότι εμείς κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και σε άλλες χώρες. Προτείνω λοιπόν να γίνει το ίδιο και στις υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης. Εάν κάποιος έχει ερωτήσεις για το δημιουργικό αυτό και πολιτιστικό κικ, την περίφημη αυτή κοινότητα που διαθέτουμε εμείς στην Αγγλία, ας έρθει σε επαφή μαζί μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχουν τίποτα να πούν οι συνάδελφοι, ναι, παρακαλώ. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι για το πώς θα το διαδώσουμε πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, εμείς φταίμε αν ζητάμε μια πρωτοβουλία για τις έξιμες πόλεις στην Ευρώπη. Προϋπολογίζουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν περιλαμβάνονται οι τοπικοί κόμβοι ή οι περιφερειακές ερευνητικέ κοινότητες. Πώς θα διαδοθούν ε, τα νέα αν δεν το κάνουμε πολύ πιο σωστά όπως κάνουμε στην επιστήμη και τη διπλωματία όπου για πρώτη φορά θα έχουμε κόμβο στο Ισραήλ που οι Ισραηλοί είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτά τα ζητήματα και στην επιχειρηματικότητα. Πώς θα διαδοθεί λοιπόν εάν ε, δεν φτιάξουμε μια γέφυρα προς το πρόγραμμα ορίζων πώς μπορούμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι εστιάζουμε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας αλλά το ερώτημα είναι σε ποιο πλαίσιο βρίσκεται και αν δεν γίνει αυτό σε άλλα έργα, ε, καμία, κανένα από τα επιχειρησιακά α, προγράμματα δεν θα ζητηθεί από, το, από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως λέμε στα κράτη-μέλη. Μπορούμε να πούμε, αν θέλετε να ζητήσετε λεφτά από τα διαρθρωτικά ταμεία, δώστε μας μια ιδέα πώς θα τα συνδυάσουμε με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Γιατί ζητάμε τα κράτη-μέλη να ξοδεύουν το 1 τρίτο των διαρθρωτικών ταμείων σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά δεν είχαμε ποτέ την ιδέα υποχρεωτικών κριτηρίων για επιχειρησιακά προγράμματα για να γίνει αυτό. Οπότε περιμένουμε με αυτό το μικρό προϋπολογισμό να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά δεν γίνεται ε, αν δεν το εντάξουμε στον ευρύτερο προϋπολογισμό που θα μας δώσει πολύ περισσότερα μέσα και μετά ελέγχουμε και λέμε «Α, είναι πολύ μικρό και δεν κάνει τίποτα». Ευχαριστώ. Ε, εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουμε τον αναπληρωτή γενικό, την αναπληρωτή γενική διευθύντρια, η κυρία Χόφμαν. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί εισηγητές, ε, συγχαρητήρια και για την εκλογή σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσετε τον λόγο και την ευκαιρία να συνοψίσω καινοτομίε και επιτεύγματα που έχουμε στην πρόταση αυτή. Οι προτάσεις αυτές για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας έχουν στόχο αφενός να ευθυγραμμίσουν το πλαίσιο του Ινστιτούτου στο μελλοντικό πρόγραμμα αυτό για ορίζοντα στην Ευρώπη και από την άλλη να βελτιώσουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας για να βασιστούμε στα ισχυρά μας ε, σημεία. Για τον κανονισμό προτείνουμε να πάμε σε επαναδιατύπωση, να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο με τον αρχικό κανονισμό του 2008, την τροποποίηση του 2013 και την τωρινή πρόταση για να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Ε, προτείναμε επίσης να είναι ουδέτερο ως προς το χρόνο για να μην τροποποιείται για κάθε νέο πι δελτα πι. Καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να εγκρίνεται μια νέα στρατηγική ατζέντα για κάθε ετή περίοδο και έτσι θα διασφαλιστεί και η απαραίτητη ευθυγράμμιση με τους στόχους του προγράμματος ε, πλαισίου που καθορίζει επίσης ε, τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους που περιλαμβάνουν ε, και τον καθορισμό στόχων για τις ε, δραστηριότητες αυτές. Λοιπόν, βασικές καινοτομίες έχουμε εδώ πέρα ισχυρά στοιχεία, την αξιολόγηση δηλαδή του EIT, η έκθεση του 2017, την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 και την δική μας αξιολόγηση. Οι βασικές καινοτομίες ε, είναι ότι αφενός έχουμε διαφάνεια, ότι θα πρέπει οι κοινότητες αυτές να εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια διαφάνειας, ειδικά στην επιλογή νέων μελών και στην κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων. Το σχέδιο χρηματοδότησης θα φέρει ένα νέο μοντέλο το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο και με την ιδέα της οικονομικής βιωσιμότητας, κάτι το οποίο βασίζεται στη μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για να τους δώσουμε κίνητρα να βρουν και άλλη χρηματοδότηση. Μετά από αυτήν την περίοδο, τη συνολική περίοδο 15 ετών, Οπότε και θα πρέπει να έχει επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα. Το EIT θα έχει την δυνατότητα υπογραφής ενός μνημονίου συνεργασίας με τις κοινότητες αυτές ε, κοινοτομίε. Για την περιφερειακή διάσταση, ναι, θα πρέπει αυτά να αποτελέσουν υποχρεωτικό μέρος ε, των στρατηγικών αυτών και η Κομισιόν πρότεινε να δεσμευτεί ένα 10% για τον σκοπό αυτόν. Όσον αφορά τώρα ε, την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας ε, των ΑΕΗ. Προτείνουμε την στήριξή τους για να μπορούν να ενταχθούν καλύτερα σε αλυσίδες και οικοσυστήματα καινοτομίας και 25% του προβλησμού για τη νέα δράση θα πρέπει να αφιερωθεί σε ιδρύματα από χώρες με χαμηλή καινοτομία. Επιλογή νέων ε, τέτοιων κοινοτήτων. Προτείνεται για το 2021 μια κοινότητα πολιτισμού, μια άλλη θα βασίζεται σε προτάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχει ορίσει το Εποπτικό Συμβούλιο. Για την ε, διοίκηση θα αυξηθεί η λογοδοσία και θα τεθούν ενισχύει η στρατηγική στόχοι, συνέργειες τώρα με το EIT και άλλα κομμάτια του μέσου ορίζοντας και τέλος αναφέρθηκε το θέμα του προσωπικού και θα έλεγα ότι έχει μπει τώρα στον κανονισμό η δυνατότητα για μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι και είμαστε βεβαίως στην διάθεσή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε και πριν ξαναδώσω το λόγο στις δύο εισηγητριές μας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Μπούζεκ, γιατί τον ξέχασα πριν, ενώ είχε μπει στον κατάλογο μιλητών. Δεν θα σας κρατήσω πολύ, θα υπογραμμίσω κάτι που είπαν οι συνάδελφοι, που έθεσαν σημαντικές ερωτήσεις προς, τις, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι εύκολο να απαντηθούν, γιατί χρειαζόμαστε λύσεις που θα εξασφαλίζουν ε, τη χρηματοδότηση βιώσιμων δραστηριοτήτων στις κοινότητες γνώσης και καινοτομία. Και η εκπαίδευση είναι καλό παράδειγμα. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη συναφής ΚΙΚ μετά το 2024. Και αν δεν μεριμνήσουμε γι' αυτό, θα θέσουμε σε κίνδυνο το τρίγωνο της γνώσης ολόκληρο. Επίσης, Συμφωνώ με τα σχόλια του συναδέλφου από το Ρηνιού. Τα περιφερειακά προγράμματα καινοτομία χρειάζονται για το μέλλον και μετά το 2024. Και ας μην ξεχνούμε ότι τρεις κοινότητες γνώση και καινοτομίας, ε, η ψηφιακή, η κλιματική και η καινοτόμος ενέργεια, είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθούν για την πρώτη 15 ετία. Θα πρέπει να κρατήσουμε αμύωτη την ευθύνη των κοινοτικών θεσμικών οργάνων για αυτές τις τρεις κοινότητες. Ευχαριστώ. Κύριε Τζάμπ, είχατε συγκεκριμένη ερώτηση. Παρακαλώ, σύντομα. Ναι, μία σύντομη ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην επίσκεψή μας στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη διαπιστώσαμε ότι οι κοινότητε γνώση και καινοτομίε για την ενέργεια, το κλίμα, τα δάση κτλ. Ε, έχουν αναφυσβήτητα αξιόλογο και αξιέπαινο έργο. Ε, άλλες είναι, απέχουν πόρο από οποιαδήποτε ε, δημοσιονομική βιωσιμότητα και το 2023 είναι πολύ κοντά. Τι σημαίνει να έχουμε μνημόνιο συνεννόηση με τι κοινότητε αυτέ, Αυτή τη διευκρίνηση θα ήθελα παρακαλώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άλλη μια σύντομη ερώτηση και μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ έχω μια, μια ερώτηση προ την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι προβλέψατε και την πιθανότητα ε, συμβάσεων εργασιακών που θα υπερβαίνουν τη δεκαετία. Τι έγινε όμω με αυτού τους πρώτους προσληφθέντες, γιατί αυτή η διάταξη δεν θα ισχύει αναδρομικά. Οπότε αυτοί οι δέκα υπάλληλοι που ξεκίνησαν από την αρχή του ΑΕΤ δεν δικαιούνται ανανέωση της εργασιακής του σύμβασης, δεν τους καλύπτεται με τη νέα πρόταση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Παρακαλώ η κυρία Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια θα ήθελα να μας απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις κοινότητες γνώσης, καινοτομίας και την δημοσιονομική τους βιωσιμότητα, ε, κάθε κοινότητα γνώσης και καινοτομίας έχει διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης και πηγές χρηματοδότησης. Εμείς τις ενθαρρύνουμε ε, και γι' αυτό προτείνουμε και το νέο μοντέλο στο νέο κανονισμό. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τις σχέσεις μεταξύ του AID και των KICS και το καθεστώ των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας μετά τη 15 αιτία. Πιστεύουμε κι εμείς ότι επενδύσεις στις ΚΙΚΣ και οι κοινοτικές επενδύσεις στις ΚΙΚΣ θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρηθούν. Και γι' αυτό προτείνουμε δυνατότητα μνημονίου συνεννόησης μεταξύ του ΕΙΤ και των κοινοτήτων γνώση και καινοτομία, ώστε να παραμείνουν αυτές οι ΚΙΚΣ στη διευρυμένη οικογένεια του ΕΙΤ. Τώρα, τι θα κάνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Θα μπορούσε να θεσπίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κοινοτήτων μετά τη λήξη της 15 ετίας. Χρήση του σήματος, συμμετοχή σε διαγωνισμούς ε, του ΑΕΤ για διασυνοριακές δραστηριότητες και άλλες ε, συναφείς υπηρεσίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα βοηθούσε να κρατήσουμε τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας στο τοπίο καινοτομίας ε, της στρατηγικής μας. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Αναλύσαμε το ζήτημα του προσωπικού και η απάντηση είναι ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει Κάτι που δεν μπορεί να λυθεί με άλλο τρόπο. Και γι' αυτό στο νέο κανονισμό προτείνουμε διόρθωση τουλάχιστον για τους νέους υπαλλήλους. Και για τα τελικά συμπεράσματα θα δώσω το λόγο στις δύο συγκεκριές μας. Πρώτα, στην κυρία Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ κύριε, Προ... κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σε σχέση με την τελευταία απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των υπαλλήλων. Νομίζω ήταν λάθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση για να αποτρέψουμε ε, αυτό το, αυτή η νομοθετική παράληψη να φέρει στο δρόμο τόσους υπαλλήλου από δική μας, από αμέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομία, συμφωνώ με την εισηγήτρια. Και σε ό,τι αφορά το κριτήριο της αριστείας, να πω ότι δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας. Μακάρι να υπάρχει αριστεία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα. Πιστεύω στην αριστεία, αλλά στην αριστεία παντού. Και αν ισχύσει το κριτήριο της αριστείας, θα είχαμε πολύ λιγότερη συγκέντρωση στο ΑΕΤ από ό,τι τώρα. Σε ό,τι αφορά τις δύο νέες κοινότητες γνώση και κοινοτομία, είμαι υπέρ αυτών, αλλά να γίνει με διαφάνεια. Και συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό καθ' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς να απαντήσω διεξοδικά. Υπάρχουν κάποιες διαστάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Το θέμα της βιωσιμότητας, για παράδειγμα, που δεν είχα αναφέρει προηγουμένως. Πολύ σημαντική η βιωσιμότητα των κοινοτήτων γνώσης και κοινοτομίας. Επίσης, οι ΚΙΚΣ είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και προσπαθούν να λύσουν τα ίδια προβλήματα, αλλά σε διαφορετικούς τομείς. Οπότε, δεν θεωρώ πρόβλημα το να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κοινότητες που διαφέρουν εξ ούτως ή άλλως. Επίσης θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και να μην αφήσουμε πίσω κάποιες κοινότητες επειδή δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Είναι αδύνατο να λειτουργούν οι κοινότητε με τον ίδιο τρόπο από τη στιγμή που προσπαθούν να διορθώσουν διαφορετικά προβλήματα. Επίση, σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό μας για την επιτυχία του ΑΙΤ και αν έχει νόημα η συνέχισή του. Ε, πότε δεν έχουμε αυθόρμητη δημιουργία καινοτομίας. Χρειάστηκαν χρόνια για να δημιουργήσουμε μια καινοτομία, για να φτάσει η καινοτομία στην οικονομία και στην κοινωνία, ε, για να φτάσουν στην οικονομία τα αποτελέσματα της έρευνας. Και το AID έχει μόνο 11 χρόνια ζωής δεν είναι πολύ νωρίς και πολύ πρόωρο να εκφέρουμε αξιολογικές κρίσεις ή να κάνουμε επικρίσεις. Είτε τα αποτελέσματα του ΕΙΤ ε, δείχνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το Ινστιτούτο. Παρόλο που ε, σίγουρα επιδέχεται βελτίωση σε πολλά σημεία και οι επιδόσεις του μπορεί να είναι καλύτερες. Οπότε είμαστε υπέρ και της συμπερίληψης περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η πλειοψηφία του ε, ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού απαρτίζεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Οπότε θα πρέπει να φυσικά να περιλάβουμε μεγάλες επιχειρήσεις ε, στις κοινότητες αλλά να μην παραγωνίζουμε και να μην ξεχνούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ισορροπία φύλου πολύ σημαντικό. Και η γεωγραφική ισορροπία που αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους σε αυτό η διαπάντηση. Γενικώ πάντως πιστεύω ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να καταλήξουμε σε ένα κανονισμό που θα ανταποκρίνεται στη λύση των προβλημάτων που ζητήσαμε, θα επικεντρώνεται περισσότερο στο ρόλο του AID και θα επιλέγει και θα υπερασπίζει αυτό το μοντέλο που ήδη έχει λειτουργήσει θετικά και μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα στο μέλλον εφόσον εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και το στηρίξουμε πολιτικά και οικονομικά για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτά και περιμένω και τις γραπτές σας τροπολογίες, ε, ενώ σημείωσα όλες τις προτάσεις σας. Είμαι βεβαίω ότι θα έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καρβαλιού, έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματίας και τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, και όλους τους ε, συναδέλφους για τις προτάσεις και είμαι σίγουρη ότι θα τα βρούμε. Μιλήσαμε όλοι για την ισορροπία, τη γεωγραφική, την ισορροπία του φύλου, μια καλύτερη ισορροπία. Και μιλήσαμε και για το τρίγωνο της γνώσης Λοιπόν, οπωσδήποτε θα τονιστεί αυτό στην έκθεση και πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Παραδείγματος χάρη για το θέμα του να παραμείνει η αριστεία ως κριτήριο πρέπει να είμαστε καινοτόμοι λοιπόν να φανταστούμε ε, ότι το τελικό αποτέλεσμα ε, το κριτηρίο αυτού θα είναι μια καλύτερη ισορροπία. Και ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό του δεύτερου της δεύτερης κοινότητας ε, και αντομίας και να έχουμε και τα κριτήρια βιωσιμότητας ε, Ναι, βάση παραδείγματο χάρη την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες προσφέρουν στις διάφορες ε, περιφέρειες. Νομίζω λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο τέτοιο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και είμαι στην διάθεσή σας για να στείλετε όλες αυτές τις ε, προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ολοκληρώσαμε εδώ την συζήτηση για το θέμα αυτό. Να σας πω το επόμενο, θέμα, το επόμενο βήμα. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης 18 ε, και 19 Μαρτίου 2020, τροπολογίες πιθανότατα 24 Μαρτίου και μετά 27 και 28 Απριλίου ψηφοφορία στην Ήτρε και θα δούμε πώς ε, θα ψηφίσει η Ολομέλεια για αυτές τις δύο εκθέσεις. Περνάμε στο σημείο υπαριθμών 12 να επιταχύνουμε αλλά θα υπάρχει και χρόνος ε, για ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν για την εφαρμογή των ε, συστημάτων δικτύων και πληροφορικής. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάνκουμ Ωρα, την τμήματάρχη της, ε, του αρμόδιου τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Connect. Ε, περιμένω τώρα να έρθει εδώ για να τα δει καλύτερα και να μας εξηγήσει την άποψη της Κομισιόν. Να σας υπενθυμίσω ότι η σχετική οδηγία εγκρίθηκε από το Κομισιόν τον Ιούλιο του 2016. Προθεσμία μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο ήταν Μάιο του 2019. Πρώτη εξέταση πρέπει να υποβληθεί 9 Μαΐου 2021. Τα κράτη-μέλη είχαν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018 να δουν ποιοι παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες όπως ηλεκτρισμό, μεταφορές ε, κτλ και ψηφιακές ε, υπηρεσίες όπως διευθύνσεις ίντερνετ και τα σχετικά και η πρώτη αυτή έκθεση εστιάζει στο πώς ε, έχουν ακριβώς τα κρατημέλη ταυτοποιήσει τις, ε, τους παρόχους αυτών των βασικών υπηρεσιών. Βρίσκουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχουν σοβαρές ασυνέπειες. Θα ήθελα τώρα ο κύριος Μπορατίνσκι να μας εξηγήσει περισσότερο αυτά τα ζητήματα και άλλες σχετικές πτυχές που αφορούν την οδηγία αυτή και θα μας μιλήσει βεβαίως. Ε, εγώ εντωμεταξύ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μιλήσετε πάνω από 10 λεπτά και οι βουλευτές μπορούν να ζητήσουν τον λόγο. Θα έχουν προτεραιότητα βεβαίω οι συντονιστές, αλλά θα έχουμε μόνο έναν γύρο παραμβάσεων για να τελειώσουμε στις 4.45. Έχετε τον λόγο κύριε Μπόρετινσκι; Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο. Η οδηγία αυτή για εμάς είναι ένας ε, πυλώνας ε, του πλαισίου ασφάλειας ένα πολύ βασικό κομμάτι της σχετικής ε, νομοθεσίας δεν ήταν κάτι το εύκολο οι διαπραγματεύσεις αυτές χρειάστηκαν τρία χρόνια Ε, για να καταλήξουμε κάπου επιτυχώς ε, και βεβαίως ε, εντάξει, σχετικά καλά τα πήγαμε. Να σας πενθυμίσω λοιπόν το εξής. Η οδηγία αφορά τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε κάποιες βασικές ικανότητες στο επίπεδο κρατών μελών. Δεύτερον, να υπάρχουν κάποιες εταιρείες στους κρίσιμους τομείς που θα έχουν κάποιες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και θα ενημερώνουν για τα σημαντικά συμβάντα και το τρίτο αφορά μηχανισμούς για συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή λοιπόν εγκρίθηκε στα μέσα του 2016 η ημερομηνία της μεταφοράς στο Εθνικό δικαίωμα ήταν ο Μάιος του 2018 η μεταφορά προφανώς ήταν δύσκολη για αρκετά κρατημέλη. Παρόλα αυτά, τελικά τον Σεπτέμβριο όλα τα κρατημέλη μας ειδοποίησαν ότι το έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Βεβαίω αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ακόμα το τι συμβαίνει, αλλά έχει επιτευχθεί ένα βασικό ορόσημο και η βασική νομοθεσία υπάρχει. Ο κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκε ακριβώς το θέμα αυτό της ταυτοποίησης των παρόχων βασικών υπηρεσιών, ένα από τα δύσκολα κομμάτια της οδηγίας και πράγματι είχαμε μια μοναδική κατάσταση είναι μια οδηγία η οποία εγκρίθηκε με βάση το άρθρο 114 εσωτερικής αγοράς. Βεβαίως, ε, ο τελικός στόχος της ε, οδηγίας, οι εν λόγω εταιρείες ε, δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης μία-μία από τα κράτη-μέλη. Οπότε υπήρχαν ανησυχίες για το θέμα αυτό. Παραδείγματος χάρη υπήρχε ζήτημα για την ομοιομορφία της εφαρμογής ε, ήδη πριν από την πλήρη έκθεση που θα συνταχθεί τον Μάιο του 2021. Τα κράτη-μέλη είχαν ακόμα 6 μήνες για να ταυτοποιήσουν τους παρόχους αυτούς, οπότε η προθεσμία ήταν Νοέμβριος του 2018. Υποτίθεται ότι θα γράφαμε την έκθεση 6 μήνες αργότερα, αλλά τελικά είχαμε όντως κάποιες ε, καθυστερήσεις, οπότε περιμένουμε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Οπότε τελικά τα καταφέραμε τέλειο Οκτωβρίου. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά στην έκθεση. Αν δείτε τα συμπεράσματα, θα δείτε ότι η έκθεση διαπιστώνει κάποια κενά στην ομοιόμορφη εφαρμογή. Ε, δηλαδή, τι εννοούμε ομοιόμορφια. Πάμε με είναι εταιρείες που λειτουργούν στον τομέα της ενέργειας, ε, των χρηματοοικονομικών ή των τραπεζών. Ε, κανονικά θα έχουν ένα παρόμοιο πεδίο και μέγεθος δραστηριοτήτων ε, θα ταυτοποιούνταν ή όχι βεβαίω αν δεν είναι σημαντικές συστημικά. Κοιτάξαμε λοιπόν τις ε, πληροφορίες ε, που λάβαμε που αφορούσε την ταυτοποίηση των σημαντικών υπηρεσιών που παρέχουν αυτές οι εταιρείες και είδαμε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το βαθμό λεπτομέρειας Οπότε, εντάξει, ε, παραδείγματος μερικέ μερικές φορές λένε απλά ότι ε, μια εταιρεία παρέχει ηλεκτρισμό. Άλλες φορές είναι πολύ πιο λεπτομέρειες ε, οι πληροφορίες λένε ας πούμε παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού κτλ. Τέλος πάντων δεν θέλω τώρα να σας πω τις λεπτομέρειες. Απλά υπάρχουν όντως κάποιες ανομοιομορφίες μετά διαπιστώσαμε κάποιο κατόφλι του χάρη ε, το πόσο ηλεκτρισμός παράγεται ε, ή συνδεδεμένα αυτόνομα συστήματα ναι, και εκεί πέρα βλέπουμε πολύ σημαντικές διαφορές πάλι οπότε υπάρχουν ε, διάφοροι βάθμοι αριθμού εταιριών που έχουν ταυτοποιηθεί ως πάροχοι σημαντικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της ε, ανάλυσης ε, είναι όταν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, αλλά ήδη από αυτή την φάση βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος κατακαιρματισμός και αυτό ίσως επηρεάσει, ξέρετε, εμέσως ε, την κυβερνοασφάλεια λόγω της ε, διασυνοριακής εξάρτησης και μπορεί να επηρεάσει και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Κάποιες χώρες ε, θα επηρεαστούν από τις ε, υποχρεώσεις που προκύπτουν σε αυτές. Αλλά εντάξει, αυτό είναι συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι ότι κοιτάμε εντατικά την εθνική εφαρμογή, οπότε εγώ με την ομάδα μου επισκεπτόμαστε όλα τα κράτη-μέλη και μέχρι στιγμής ε, έχουμε μιλήσει με τις αρχές. Ε, σε κάποιες χώρες, τις λιγότερες, υπάρχει μια κεντρική αρχή και τέλος. Αλλού είναι αποκεντρωμένες οι αρμοδιότητες. Και βεβαίω ε, μιλάμε και με συνομιλητές μας στις ε, κυβερνήσεις, οπότε έχουμε ένα πολύ καλό δείγμα και εταιριών και επαγγελματικά πρέπει να πω είναι κάτι το πολύ ικανοποιητικό γιατί βλέπουμε να έχουμε συχνά πραγματικό αντίκτυπο. Και χάρη στην οδηγία αυτή, παραδείγματος χάρη, είχαμε την δυνατότητα να απασχολήσουμε τέσσερις φορές περισσότερους ειδικούς στα ζητήματα αυτά στην κεντρική αρχή σε ένα κράτος μέλος. Ε, σε ένα άλλο κράτος μέλος μίλησα με άτομα στο επίπεδο της εταιρεία που μας είπαν ότι με την εφαρμογή της εταιρεία ε, τους παίρνει για πρώτη φορά στα σοβαρά το Διοικητικό Συμβούλιο. Οπότε βλέπουμε αυτό να υπάρχει και βλέπουμε προφανώς ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Υπάρχουν χώρες που πρέπει να υιοθετήσουν ε, επιπλέον ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, και παρά το ότι ήταν 2016 νομίζω ότι είμαστε σε μια αρκετά πρώτη φάση, πρώιμη φάση της εφαρμογής της οδηγίας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, η προθεσμία για την αναθεώρηση είναι το Μάιο του 2021. Παραδείγματος χάρη ε, ο Επίτροπος Λεμπερτών είπε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2021. Τέλος. θα έλεγα ότι έχει συσταθεί ακριβώ αυτό ο φορέα που προβλέπει η οδηγία. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Μαζεύονται τα κράτη-μέλη να συζητήσουν τι εμπειρίε τη και πρόκειται για τον βασικό φορέα που συντονίζει τι προσπάθειε των κρατών μελών πέρα από την εφαρμογή τη οδηγία. Και ίσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δουλειά που έγινε προσφάτω για την ασφάλεια των δικτύων πέμπτη γενιά, το οποίο είχαμε ακριβώ εμπιστευτεί στην ομάδα αυτή, την οποία στήριξε η Κομισιόν. Η ΕΝΙΣΑ επίσης με τη νέα της ε, εντολή ε, με το νέο νομοθέτημα παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών. Οπότε θα έλεγα ότι προχωράμε με νέες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι η πλήρης εφαρμογή είναι το, το βασικό και πραγματικά αξίζει και πόρους αλλά και την πολιτική προσοχή του ε, Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας και διότι σεβαστήκατε το χρόνο που είχαμε. Έχω ε, δύο αιτήματα εκ μέρους των συναδέλφων για να λάβω το λόγο. Αν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος, εάν τους εμπνεύσουν αυτές οι δύο πρώτες ερωτήσεις που θα τεθούν, θα δώσω το λόγο. Αρχίζω με την κυρία Πιλάρδα Καστίγιο. Το μικρόφωνο παρακαλούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι μάθαμε όλοι που βρίσκεται το περίφημο νης και που βρίσκονται οι εξελίξεις. Μας εξηγήσατε κάποια πράγματα. Είναι απολύτως σαφές Σύμφωνα με αυτά που είπατε και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ε, ε μεθοδολογίες, έχουν δώσει διαφορετική ερμηνεία στο τι είναι μια βασική υπηρεσία και γι' αυτό υπάρχει και ο κατακαιρματισμός που είναι εντελώς αντίθετο ε, από τον στόχο αυτής της οδηγίας. Εάν έχουν έτσι λοιπόν τα πράγματα, η, αναδιο... αναδιάρθρωση, οι αλλαγές της οδηγίας νης για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων κρατών μελών για αυτά τα θέματα είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς απαραίτητο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. δεδομένου ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και επί αυτού θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερα να σκεφτούμε περισσότερο μήπως πρέπει να έχουμε κανονισμό για οδηγία, διότι εκεί έχουμε πάρα πολύ με ευρύ πεδίο ερμηνείας σε έναν τομέα στον οποίο είναι εντελώς απαραίτητο να έχουμε σαφή τρόπο ερμήνευσης κάποιων γεγονότων και το συντομότερο δυνατό, όχι να μακρύ. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν ενδιαφέρον και πάρα πολύ καλό η όλη αναθεώρηση και οι να οδηγήσουν σε κανονισμό παρά σε οδηγία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Δελκαστήλιο. Κύριε Κριστόφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι τζάμπο στην ε, Βουλγαρία υπέστη μία κυβερνοεπίθεση και έτσι τα προσωπικά δεδομένα πάρα πολλών χιλιάδων χρηστών δημοσιοποιήθηκαν. Στα πλαίσια των επισκέψεων της Επιτροπής, θα ήθελα να ρωτήσω, έχει πάει ε, στην Βουλγαρία για να ερευνήσει τέτοιου είδου θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ναι, ποια είναι η εντύπωση που σας δημιουργήσε. Ευχαριστώ κυρία Βερκούνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να πω το εξή. Όταν μιλούμε για κυβερνοασφάλεια, εννοούμε ότι πρέπει να παίρνουμε μέτρα σε όλα τα επίπεδα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο επιχειρήσεων, εσείς πού πιστεύετε ότι υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, πού θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα στην κοινωνία, στις ε, ε, καθημερινότητά μας, στις επιχειρήσεις, μήπως δεν έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας αρκετά στην κυβερνοασφάλεια ε, σε κάποια επίπεδα, σε κάποιες χώρες περισσότερο πόλο, σε κάποιες επιχειρήσεις, σε επίπεδο ε, τοπικής ε, αυτοδιοίκησης, σε κάποιες τεχνολογίες στις οποίες ξέρουμε ότι υπάρχουν σήμερα ε, κάποιοι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας. Πιστεύετε ότι κάνουμε αρκετή κατάρτιση και αρκετούς ελέγχους στα κράτη-μέλη επίσης και στις διάφορες οργανώσεις τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουμε κατάλληλα και να καταρτήσουμε τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τέτοιου θέματα, διότι υπάρχουν κίνδυνοι. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και δεν ζητά κανένας συνάδελφος το λόγο, θα σας παρακαλέσω παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και κάποιες ε, ε παρατηρήσεις ολοκληρώνοντας. Ο κύριος Κλάουσμπουργκερ όμως βλέπω ότι ζητά το λόγο. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι με είδατε. Έχουμε δύο διαφορετικά θέματα εδώ και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρώτα απ' όλα, ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο κάποια δεδομένα μπορούν να δοθούν σε κάποιον τρίτο και υπάρχει και ο παράνομος, ο παράτυπος. Το δεύτερο, ο παράτυπος τρόπος, νομίζω ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς από μια τέτοιου είδους οδηγία, δεδομένου ότι είναι παράνομη δραστηριότητα αυτή. Οι δυνατότητες που προσφέρονται για να ε, μπορέσει κανείς να μπει στα δεδομένα ε, κάποιου για να κάνει κάποιες συναλλαγές με παράνομο τρόπο είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλες. Στην Ευρώπη έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο ε, μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα παράνομα και οι κυβερνήσεις παρά το γνωρίζουν δεν κάνουν τίποτα για να καταπολεμήσουν ως φαινόμενο. Θα είναι λοιπόν να αρχίσουμε τη συζήτηση από εδώ ένας καλός τρόπος. Θα πρέπει όμως να σταματήσουμε τις παράνομες ε, μεταφορές και διαβιβάσεις δεδομένων που συμβαίνουν παντού στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Να ευχαριστήσω κυρία, την κυρία Ντελκαστήγιο πρώτα για τα σχόλιά της. Ήταν πολύ υποστηρικτική στις προσπάθειές μας και στην οδηγία και στην νομοθετική πρόταση για την κυβερνοασφάλεια. Ε, φυσικά προς το παρόν όλα είναι ανοιχτά και θα αναλύσουμε τους διάφορους τρόπους ε, για να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση όπου χρειάζεται. Πάντως τα κράτη-μέλη έκαναν κάποια προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά για ήπια μέτρα. Ε, η ομάδα συνεργασία υιοθέτησε κάτι κατευθυντήριε γραμμέ για μέτρα ασφάλεια, για ειδοποίηση, για κάποια περιστατικά. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτή τη συνεργασία. Πάντω έχουμε τους παρέχοντες υπηρεσίες νέφους, για παράδειγμα, και έχουμε μία ευθυγράμμιση. Αλλά έχουμε μία ήπια προσέγγιση και μία ήπια εποπτεία που δεν είναι αρκετά ισχυρή. Ε, αντίστοιχη με αυτή των βασικών υπηρεσιών. Πάντως ε, θα έχουμε εκτενείς διαβουλεύσεις και φυσικά θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία. έχουμε επίγνωση αυτού του σημαντικού συμβάντος. Είχαμε επαφές με τις βουλγαρικές αρχές και μέσω του δικτύου EU-CERT που είναι η μονάδα ανταπόκρισης περιστατικών σε υπολογιστές ε, είναι δίκτυο που παρέχει μια βοήθεια για τα θέματα αυτά και ειδοποιηθήκαμε Έχουμε επισκεφτεί και τη Βουλγαρία, αλλά σε αυτή τη φάση τη διαδικασία δεν μπορούμε να σα ενημερώσουμε για τα πορίσματά μα. Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο τη έρευνα. Και σίγουρα η έκθεσή μα θα έχει πιο γενικό χαρακτήρα. Λυπάμαι, αλλά σε αυτή τη φάση δεν είμαι σε θέση να σας ενημερώσω πιο αναλυτικά. Σίγουρα έχουμε διαφορετικά, διαφορετικά στάδια ορίμασης στα κράτη-μέλη ως προς την οδηγία. Και γι' αυτό θεσπίσαμε και την οδηγία που έχει περισσότερο νόημα για τις χώρες που υστερούν κάπως. Και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το πρόγραμμα εργασιών, για τη συνεργασία, και αυτή ήταν η ιδέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, πιο απτή και μέσω των ετησίων προγραμμάτων μπορεί και να ε, παρακολουθεί. Έχουμε ε, και το έρασμος για ανταλλαγές ε, εμπειρογνωμόνων κυβερνοασφάλειας και έχουμε κάποιο μικρό κονδύλιο για να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα του χρόνου. Επίσης υπάρχει μια πρόταση για αξιολογήσεις ομοτήμων Στην πορεία θα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά, κάτι που δεν είναι εύκολο, γιατί σίγουρα η κυβερνοασφάλεια εφάπτει σε κάποια σημεία με την εθνική ασφάλεια. Οπότε δεν μπορούν όλα να είναι αντικείμενο ανοιχτής πανευρωπαϊκής συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική σας ερώτηση, ε, το εγχείρημα της οδηγίας νης μας δείχνει ότι είναι σε διαφορετική φάση και οι τομείς και τα κράτη-μέλη, διαφορετική φάση ορίμασης. Σε ό,τι φορά την παρακολούθηση των κινδύνων και δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις εύκολα. Σε μερικούς κλάδους ε, ο κίνδυνος εμφανίστηκε σε πρώιμο στάδιο και οδήγησε σε σημαντικές ζημίες, κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Να δούμε τις ε, διάφορους κλάδους, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχουμε τη μεγαλύτερη ορίμαση των αμ, το, της άμυνας σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Και έχουμε και πολλές δραστηριότητες ε, πανευρωπαϊκές, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και στα κράτη-μέλη, όταν μιλούμε με εμπειρογνώμονες της κυβερνοασφάλειας της τράπεζας, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο προηγμένοι από τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες άλλων τομέων. Ε, άλλος ε, κλάδος, στον οποίο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στην κυβερνοασφάλεια, είναι τα νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία επεξεργάζονται τεράστιο αριθμό στοιχείων δεδομένων, προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Επίσης, αυξάνεται η ελεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών ε, και των διαφόρων επιχειρήσεων και εγχειρήσεων που γίνονται στα νοσοκομεία. Και όλα αυτά είναι τμήματα της υποδομής και εκεί πολλά θα πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η κυβερνοασφάλεια. Πάντως τα νοσοκομεία εξορισμού δεν είναι τόσο εύπορο όσο οι τράπεζες. Και γι' αυτό θα πρέπει το σημείο αυτό να το αναλύσουμε ιδιαίτερως. Οι δημόσιες διοικήσεις δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή οδηγία. Αρχικά προβλεπόταν στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη. Αυτό που εκαναν όμω όμως πολλά κράτη-μέλη κατά τη μεταφορά τη οδηγία στο εθνικό του δίκαιο είναι να το συμπεριλάβουν, αλλά αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Πάντω τα κράτη-μέλη λαμβάνουν εθνικώ κάποια μέτρα για να προστατεύσουν ε, τις δημόσιες διοικήσεις τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για τι άλλε τεχνολογίες, αυτόνομη, αυτοματοποιημένη οδήγηση, τεχνητή νοημοσύνη, 5G, πέμπτη γενιά κινητών, επίση κυβερνό σε όλους αυτούς τους τομείς η κυβερνοασφάλεια είναι σημαντικό τμήμα της λύσης και σημαντικό στοιχείο των τεχνολογιών. Σε ό,τι αφορά την τελευταία ερώτηση, δεν γνωρίζω. Πάντως αυτό που μπορούμε να κάνουμε με την οδηγία της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι να δημιουργήσουμε αθεκτικότητα σε θέματα κυβερνοασφάλειας, να δημιουργήσουμε άμυνες και τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις, οι δημόσιες διοικήσεις και οι διάφορες οργανώσεις να προστατευτούν καλύτερα από κυβερνοεπιθέσεις. Μερικές φορές μια ΜΜΕ ακούμε πολλά για κυβερνοεπιθέσεις. Η οδηγία όμως νης ε, περιλαμβάνει και άλλους κινδύνους. Και έχουμε πολύ σημαντικά συμβάντα που δεν είναι αποτέλεσμα κακόβουλων ε, δραστών. Έχουμε θέματα ε, ελέγχου της ενέργειας κυκλοφορίας που ε, επλήγησαν από κάποιο συμβάν τέτοιο λόγω κακής ενημέρωσης του λογισμικού τους. Δεν ήταν ε, κάποιο συμβάν αποτέλεσμα κατά ανάγκη κακόβουλης ενέργειας. Επίσης έχουμε και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Αυτό όμως εντάσσεται σε ξεχωριστό νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο και η παράνομη ε, ε, παρεμβολή είναι ένα από τα βασικά εγκλήματα. Επίσης, πρόκειται, έχουμε και την οδηγία του 2011 για την επίθεση στα συστήματα πληροφοριών που θα αναθεωρηθεί και αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα των προληπτικών δράσεων για τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τα σχόλιά σας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών και προσπαθούμε όσο μπορούμε να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση αλλά και να ενισχύσουμε την ικανότητα στη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Και για τις κρίσιμες υποδομές το θέμα της κυβερνοασφάλειας λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ε, ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσει, προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές και φυσικά να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρέμειναν μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίας της Επιτροπής μας. Μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας τώρα της δημόσιας μας συνεδρίασης και θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 5 που θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Οι υπόλοιποι ραντεβού αύριο το πρωί με την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Ενέργειας αύριο στις 9 η συνέχεια της δημόσιας συνεδρίασης. Ευχαριστώ. καλός σας απόγευμα.